σχετικά έγγραφα. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Κοέγιο. Για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μπαρό, αξιότιμοι βουλευτές. Αυτό που σήμερα συζητούμε έχει ε, ως στόχο την αναθεώρηση του κανονισμού 2004 που έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα βιομετρικά στοιχεία στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας και την εισαγωγή ε, βιομετρικών στοιχείων. Τώρα είμαστε στη συναπόφαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γαλλική Προεδρία και τον Επίτροπο κύριο Μπαρό για την επιμέλεια που έδειξαν για να καταλήξουμε σε πρώτη ανάγνωση. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις ηγητές που βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Είναι τελείω απαραίτητος αυτός ο κανονισμός. Το 2004 άρχισε να ισχύει και από τον Ιούνιο και μετά όλα τα κράτη-μελή ήταν υποχρεωμένα να συλλέγουν στοιχεία για τα παιδιά. Γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις σε διάφορα κράτη-μέλη. Είναι πολύ δύσκολο όμως να ε, συλλέγονται στοιχεία ε, τέτοια βιομετρικά για παιδιά κάτω των 6 ετών. Βέβαια μπορούν πάντα να υπάρχουν ε, εξαιρέσεις σε αυτή την υποχρέωση. Αυτό σημαίνει μόνο ότι ε, στην περίπτωση αυτή εκδίδονται προσωρινά και μόνο διαβατήρια και αυτό είναι οικονομική επιβάρηση αλλά και γενικότερα για τους γονείς. Κάθε φορά που πρέπει να ταξιδέψουμε το παιδί τους να ζητούν καινούριο διαβατήριο. Μετά από τέσσερα χρόνια καταλήψαμε τα έξι έτη και μιλούμε για παιδιά άνω των 12 ετών. Υπάρχει και ρήτρα αναθεώρηση μετά το πέρα τη τετραετία και λαμβάνοντα υπόψη τη μελέτη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε. το σύστημα και ποια είναι η αξιοπιστία αυτών των στοιχείων και από εκεί και πέρα θα εναρμονιστεί ε, το όριο ηλικίας για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και δεύτερη εξαίρεση για τα πρόσωπα εκείνα που για διάφορους λόγους ε, είναι σε ε, αδυναμία σωματική να δώσουν αυτά τα αποτυπώματα. One person, one passport. Επίσης υπάρχει σύσταση του ΙΚΑΟ. Δηλαδή ένα διαβατήριο αναπρόσωπο, καθένας να είναι κάτοχος ενός και μόνο διαβατηρίου. Αυτό είναι επιπλέον ε, πλεονέκτημα και μας βοηθάει στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών και του τράφικινγκ. Θα πρέπει να υπάρχει και μια κοινή θέση των θεσμικών οργάνων για την προστασία των ανηλίκων για κοινού κανόνες αναρμονισμένους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει, θα προτείνει μάλλον διάφορα μέτρα. Εμείς βέβαια δεν έχουμε εκεί πολλές ε, αρμοδιότητες, διότι τα διαβατήρια εμπίπτουν στις ε, κρατικές αρχές που τα εκδίδουν. Η Ευρώπη το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ισχύει τα βιομετρικά στοιχεία που είναι υποχρεωμένα να αναγράφονται στα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη διέλευση συνόρων. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει στη θέσπιση κανόνων που έχουν να κάνουν με τη διάσταση των φωτογραφιών και άλλα τεχνικά στοιχεία. Είναι συγκεκριμένος ο κανονισμός, συγκεκριμένοι οι κανόνες και τα έγγραφα που χρειάζονται για τη διέλευση των συνόρων. Για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας, για να καταλάβουμε αν ο κάτοχος πραγματικά είναι ο γνήσιος κάτοχος εκείνος που ταξιδεύει. Επίσης, ε, κατά τη διέλευση των συνόρων, θέλουμε να ε, καταπολεμήσουμε και το έγκλημα, αλλά και να μην έχουμε ψευδείς δείκτες ε, άνησης και απόρριψης. Υπάρχει και έννοια του Ευρωπαίου επόπτη προστασία των ανηλίκων και των στοιχείων δεν ελήφθη όμω υπόψη κατά την εκπόνηση αυτή τη πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Κόγιο. Εξ ονόμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο έχει κύριο Μπαρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, τον Κάρλος Κοέλιο, για την εξαίρετη εκθεσή του και επίσης για την εξαίρετη συνεργασία με την Επιτροπή πάνω σε ένα θέμα λεπτό και ευαίσθητο. Η πρόταση της Κομισιόν απέβλεπε στην εισαγωγή εναρμονισμένων εξαιρέσεων στην απέτηση συλλογής των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ούτως ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να την χάνουν της ίδιας μεταχείρισης. Εκτός αυτού η Κομισιόν ήθελε να προστατεύσει τα παιδιά από την, το λαθρεμπόριο των παιδιών βάσει της αρχής που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, δηλαδή ένα άτομο, ένα διαβατήριο. Θα ήθελα να χαιρετήσω τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση στο μέτρο όπου τα δακτυλικά αποτυπώματα πρέπει να ενσωματώνονται στα διαβατήρια το αργότερο στις 28 Ιουνίου 2009 εάν μια συμφωνία δεν βρεθεί όλοι θα ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα ακόμα ε, και τα παιδιά που μόλις γεννηθούν εφόσον πρέπει να ταξιδεύουν με ένα διαβατήριο. Θέλω λοιπόν να εκφράσω την ικανοποίηση της Κομισιόν για την διαπραγματευμένη πρόταση συμβιβασμού. Τώρα η Επιτροπή θα ασχοληθεί με την έκθεση που ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μακρηγορήσω. Θα ακούσω τώρα με ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ όμως άλλη μια φορά τον εισήγησή σας, τον κύριο Κάρλος Κοέλιο που έκανε μια εξαίρετη εργασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Γκάσεκ. Mr President, dear colleagues, I am happy on behalf of the EPP to support the proposal. μεγάλη μου ικανοποίηση υποστηρίζω τις προτάσεις που ε, υποβλήθηκαν σήμερα εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι απαραίτητο να υπάρξουν κοινέ προδιαγραφές για την επαλήθευση των βιομετρικών δεδομένων. Υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις και ίσως να μην το γνωρίζουν οι συνάδελφοί μου αυτό σχετικά με το πόσο ε, προσεκτικά επαληθεύουν τις φωτογραφίες των διαβατηρίων. Πολλές χώρες ζητούν να ε, λαμβάνονται φωτογραφίες των ε, προσώπων και ε, απαιτούν ο ίδιος ενδιαφερόμενος να εμφανιστεί με τη φωτογραφία του ενώπιον του ε, υπαλλήλου που εκδίδει το διαβατήριο. Όμως, αλλού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτά γίνονται δια του ταχυδρομείου και η αυθεντικότητα της φωτογραφίας γίνεται από έναν λεγόμενο επαγγελματία, ο οποίος οφείλει να γνωρίζει το πρόσωπο τουλάχιστον μία διετία. Ο κατάλογος των προσώπων που έχουν το δικαίωμα να το πράξουν αυτό είναι πραγματικά ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορεί να το κάνει ο οδοντίατρός σας ή ο πτωμέτρης σας ή και ένας επαγγελματίας φωτογράφος. Και βεβαίω ε, με όλο το σεβασμό που έχω για τα μέλη των επαγγελμάτων αυτών. Είναι λοιπόν πολύ χαλαρή η ρόλη επαλήθευση και το ίδιο και στι ΗΠΑ Η επαλήθευση των φωτογραφιών για τα διαβατήρια, για όσου για πρώτη φορά αποκτούν διαβατήριο, μπορούν να γίνουν σε κατάλληλα οικήματα. Δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει και στο τοπικό ταχυδρομείο φαίνεται να είναι ε, πραγματικά απίστευτο για μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες ε, ε, ενδιαφέρονται και ανησυχούν τόσο πολύ για την ασφάλεια και όπου οι Αμερικανοί υπήκοοι δεν χρειάζονται για παράδειγμα βίζα για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν να είναι πιο αξιόπιστα τα βιομετρικά δεδομένα και εννοώ τα δακτυλικά αποτυπώματα αλλά και οι αρχές που επαληθεύουν, που ελέγχουν τα διαβατήρια πρέπει να έχουν κοινέ προδιαγραφές και ιδίως οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όπου ε, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα αλλά και οι ε, κάτοικοι των ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάσεκ. Το λόγο τώρα έχει εξ ονόματος σοσιαλιστών για δύο λεπτά η κυρία Ρουρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά την υιοθέτηση του 2004 του κανονισμού για τα πρότυπα για την ασφάλεια και την ενσωμάτωση των βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια, τα κράτη-μέλη δεν είχαν προβλέψει καμία εξαίρεση για την συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τώρα, αποτυπωμάτων. Τώρα μα βλέπουμε ότι η τεχνολογία δεν εξασφαλίζει τα δακτυλικά αποτυπώματα των ε, παιδιών κάτω των δύο ετών να είναι αρκετά αξιόπιστα για να χρησιμεύσουν για την ασφάλεια ε, στα διαβατήρια. Χαίρομαι ε, για τον συμβιβασμό σχετικά για την συλλογή των βιομετρικών στοιχείων με ρήτρα αναθεώρησης σε τρία χρόνια. Εμείς ε, δεχτήκαμε την εξαίρεση για τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη μια νομοθεσία. Η χρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων γίνεται αποδεκτή μόνο αν επιτρέπει να προστατεύσουμε πράγματι τα παιδιά μας. Αυτή δεν είναι η περίπτωση και είμαστε ανοιχτοί σε μια ενδεχόμενη θετική εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Η προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των παιδιών που ταξιδεύουν μόνα τους, ούτως ώστε να προλάβουμε κάθε απαγωγή ε, ή κάθε εμπόριο παιδιών. Η ενσωμάτωση των βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια των παιδιών δίνει μια εσφαλμένη εντύπωση ασφαλείας, διότι δεν εμποδίζει ένα παιδί να διασχίσει ένα σύνορο χωρίς την άδεια των γονέων. Ο συμβιβασμός με τα κρατημέλη θα επιτρέψει στην Επιτροπή να παρουσιάσει μια έκθεση για τις απαιτήσει για τους ανήλικες που ταξιδεύουν μόνοι τους αυτή η έκθεση θα μας επιτρέψει να, να, να προτείνουμε πρωτοβουλίες για να εγγυηθούμε μια ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση. Τα στοιχεία, τα βιομετρικά των διαβατηρίων πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ε, για να εξεκριβωθεί η γνησιότητα του εγγράφου και η χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων ευαισθητών όπως είναι τα βιομετρικά στοιχεία και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αυστηρούς κανόνες προστασίας των προσωσικών δεδομένων. Ευχαριστώ την κυρία ε, Ρουρ. Δύο λεπτά. Ο κύριος Ντεπρέ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισήγη μας τον Κάρλος Κοέλιο και την πρώην Γαλλική Προεδρία που δεν είναι παρούσα. Είναι φυσικό διό για την συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση χρειαζόταν η βούληση και χρειαζόταν η ικανότητα να συμφωνήσουμε για τους απαιτούμενους συμβιβασμούς. Ε, ευχαριστώ τον Κάρλος ε, διότι η αιτιολογική σκέψη είναι ένα μικρό θαύμα ε, ε, ευφυΐας και διεξοτεχνίας πολιτικής. Αν αναλύσουμε το κείμενο το οποίο μας προτείνεται, Υπάρχει μια μεγάλη αρχή που είναι η επαναστατική αρχή αυτής της έκθεσης. Δεν είναι τα βιομετρικά στοιχεία που είχαν αποφασιστεί από το 2004. Είναι η αρχή ένα άτομο, ένα διαβατήριο. Ε, πράγμα που θέτει το πρόβλημα των παιδιών και την ηλικία από την οποία μπορεί κανείς να παίρνει, να συλλέγει τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών. Είναι δύσκολος αυτός ο συμβιβασμός που ορισμένοι θέλαν το νωρίτερο δυνατόν για να προστατευτούν τα παιδιά όσο το δυνατόν νωρίτερα σε μικρή ηλικία, αλλά έπρεπε να έχουμε βιομετρικά στοιχεία, αξιόπιστα πράγμα που δεν είναι εξασφαλισμένο για την ώρα. Ο συμβιβασμό που έλαβε χώρα δακτυλικά αποτυπώματα είναι υποχρεωτικά από την ηλικία των 12 ετών. Τα κράτη που στα συλλέγουν νωρίτερα θα μπορούν να εξοκολουθήσουν να το πράττουν για τέσσερα χρόνια, αλλά όχι περισσότερο και θα πρέπει να αξιολογήσει η Κομισιόν το σύστημα και προτείνοντας τροποποιήσεις αν παρίσταται ανάγκη. Πρέπει λοιπόν να ελπίζουμε ότι η τεχνολογία θα κάνει σημαντικές πρόοδους διότι το ιδανικό για να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά θα ήταν να έχουμε βιομετρικά στοιχεία αξιόπιστα, συγκρίσιμα των νωρίτερο δυνατόν. Και με το πνεύμα το μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε με το κείμενο αυτό ε, που χαιρετίζω, που επικροτώ τον εισηγητή, την Επιτροπή για την αρχική της πρόταση και το Συμβούλιο ε, για το πνεύμα στο συμβιβαστικό το οποίο επέδειξε. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ για την Ευρώπη των Εθνών, την ομάδα της Ευρώπης των Εθνών. Για δύο λεπτά δίνω τον λόγο στην κυρία Αντζελίλη. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαίρετη εργασία του και ε, για ε, τα δικαιώματα των ανηλίκων. Είμαι στην Επιτροπή για τα δικαιώματα και θα ήθελα να αναφέρω, όπως και άλλοι ε, συνάδελφοι, ορισμένα σημεία της έκθεσης. Υπάρχει η αρχή της εξασφάλισης κοινών κανόνων για την προστασία των παιδιών που διασχίζουν ε, τα εξωτερικά σύνορα και ε, το, η αρχή ένα άτομο, μια, ένα διαβατήριο. Αυτό είναι, σημαντικό, ε, σημαντική αρχή διότι συνδέει τα στοιχεία με το άτομο που κατέχει αυτό το έγγραφο. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται τώρα δεν είναι απαραίτητες διότι αυτές πρέπει να έχουν την ταυτότητα του παιδιού στο διαβατήριο των γονέων και έτσι ο έλεγχος για την ταυτότητα του παιδιού είναι ε, λιγότερο αξιόπιστος και διευκολύνει τις απαγωγές ανηλίκων και την εκμετάλλευση των παιδιών. Τρίτον, η εισήγηση αυτή προβλέπει η Επιτροπή, η Κομισιό να παρουσιάσει μια έκθεση που θα αναφέρεται στην δυνατότητα, την τεχνική χρησιμοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών κάτω των 12 ετών για να μπορέσει να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους. Θα πρέπει να δούμε αν είναι αξιόπιστο το σύστημα αυτό για την προστασία των ανηλίκων. Για να κλείσω θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο στο μέλλον να προσδιορίσουμε πιο ε, προχωρημένα τεχνικά μέσα, πιο ασφαλή, ούτω ώστε να προσδιορίσουμε με βέβαιο τρόπο την ταυτότητα και την ηλικία του παιδιού και αυτό το όσο το δυνατόν πιο νωρίς ή δυνατόν από τη γέννηση. Ευχαριστώ κυρία Τζελίλη για την ομάδα των Πρασίνων και για δύο λεπτά η κυρία Σντανόκα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Εξ ονόματος των Πρασίνων θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κοέλιο για την θαυμάσια εκθεσή του. Έχουμε τις διάφορες πολιτικές μας απόψεις, αλλά ο κ. Κοέλιο κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να συμβιβάσει τις απόψεις αυτές. Εμείς έχουμε επιφυλάξει όσον αφορά τη χρήση των βιομετρικών δεδομένων μέχρι ότου αποδειχθεί η αξία τους χωρίς αμφιβολία θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να είναι εγγυημένα τα προσωπικά δεδομένα. Και σε ό,τι αφορά τη χρήση βιομετρικών δεδομένων σε προξενικές θεωρήσεις είμαστε αντίθετοι, αλλά και σε διαβατήρια. Θεωρούμε την παρούσα πρόταση ως δυνατότητα και να βάλουμε όρια στο που θα λαμβάνονται δεκτυρικά αποτυπώματα των ανθρώπων που επιθυμούν να ε, ταξιδέψουν το όριο ηλικία 12 ετών για τι ε, χώρε μέλη εκείνε όπου δεν λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών και το όριο ηλικία των 6 ετών που θεσπίζεται για τι υπόλοιπε χώρε μέλη. Θέλω να τονίσω και πάλι την υποστήριξή μα για τα όρια ηλικία, η οποία υποστήριξη δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε γενικά την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εμεί πιστεύουμε ότι τα βιομετρικά δεδομένα στα διαβατήρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την ε, επαλήθευση της γνησιότητας του εγγράφου και της ε, ε, ταυτότητας του κατόχου. Η χρήση για άλλους λόγους, όπως για την επιβολή του νόμου, δεν νομιμοποιείται ούτε υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Δεν θέλουμε να φτάσει ο κάτοχο του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου να θεωρείται συνήθι ύποπτο, του οποίου τα δακτυλικά ε, αποτυπώματα πρέπει να τηρούνται σε αρχεία. Τονίζω και πάλι ότι ε, συγχαίρουμε τον κύριο Κουέλγιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τον συμβιβασμό. Εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ενία Αριστερά, για δύο λεπτά η κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι υπέρ της ιδέας να λαμβάνονται δακτυρικά αποτυπώματα των μικρών παιδιών και μάλιστα και των μωρών. Τα παιδιά πρέπει να ξερούνται από την υποχρέωση δακτυρικών αποτυπωμάτων στα διαβατήρια. Είναι λοιπόν σωστό να υπάρξουν εξαιρέσει για τα παιδιά. Για την χρήση των βιομετρικών δακτυλικών αποτυπωμάτων για παιδιά κάτω των 12 ετών δεν υπάρχουν ακόμα ασφαλείς ε, γνώσεις. Δεν είναι και βέβαιον κατά πόσον τα δακτυλικά αποτυπώματα μικρών παιδιών που βρίσκονται στην ανάπτυξη διατηρούνται ίδια και για πόσο διάστημα. Ας ε, ε, μην φτάσουμε λοιπόν σε μικρότερη ασφάλεια από αυτήν που επιθυμούμε. Πρέπει ε, λοιπόν να τηρούνται βιομετρικά δεδομένα τα οποία να μην μπορούν να αμφισβητηθούν. Ο συμβασμός απηχεί τι επιφυλάξει αυτέ, πράγματι. Και λόγω τη επιμονή του Κοινοβουλίου και τη καλή εργασία του εισηγητού έχει ε, υιοθετηθεί το όριο των 12, της ηλικίας των 12 ετών για μια τετραετία, ώστε να μπορέσει να γίνει μια μεγάλη έρευνα για να διαπιστωθεί πόσο αξιόπιστα είναι τα βιομετρικά δεδομένα των παιδιών. Δυστυχώ όμω ο συμβασμό προβλέπει και δυνατότητα εξαιρέσεω υπερχορών οι οποίε ήδη δια νόμου έχουν θεσπίσει την λήψη δαχτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών κάτω των 12 ετών. Είναι σημαντικό λοιπόν στα πλαίσια του, του συμβιβασμού να διαπιστωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για βιομετρικά δεδομένα σε διαβατήρια και άλλα έγγραφα ταξιδιού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για να δημιουργηθούν τράπεζες δεδομένων με τέτοια δεδομένα σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κάφμαν. Ανεξαρτησία και δημοκρατία. Για δύο λεπτά ο κύριος Πάτεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευτυχώ το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρείται από τον κανονισμό αυτό αφού δεν εντάσσεται στην ζώνη Σέγγεν. Είπε όμω η Βρετανική κυβέρνηση ότι θα κάνει προσπάθειες να συμβαδίζει με την ε, ρύθμιση αυτή ώστε να μην είναι οι Βρετανοί πολίτε δεύτερη κατηγορία. Άρα δηλαδή εννοεί ότι αυτή η νομοθετική πρόταση είναι πρώτη κατηγορία. Όμω όπω δείχνει η έκθεση, τίθενται πολλά θέματα σχετικά με τη γνησιότητα των βιομετρικών δεδομένων και τη δυνατότητα επαλήθευσή του. Ποια έγγραφα χρησιμοποιούνται ω βάση για ε, την ε, υποβολή αίτηση ε, για το διαβατήριο του ενδιαφερομένου. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, έχει εκδοθεί ένα διαβατήριο, δεν είναι και πολύ χρήσιμο εάν δεν μπορεί ε, να διαπιστωθεί ταυτόχρονα και η ταυτότητα του κατόχου με κάποιον άλλο τρόπο και σε βάση μιας άλλης ε, τράπεζας δεδομένων. Η έκθεση λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς τρόποι διατήρησης των δεδομένων αυτών, αλλά από την εμπειρία μας στη Βρετανία γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Προσωπικές πληροφορίες ε, υψηλής ευαισθησίας εκατομμυρίων ανθρώπων χάθηκαν τα τελευταία χρόνια από ε, αμέλεια της κυβέρνησης στην Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι γνωρίζουν πλέον ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι ασφαλή στα χέρια της Βρετανικής κυβέρνησης. Δεν μιλεί η έκθεση και για τις σχετικές ευθύνες. Η δοκιμαστική περίοδος που έγινε το 2004 έδειξε μεγάλη πιθανότητα σφαλμάτων και ε, για ε, ε, την ηλεκτρονική αναγνώριση και στη βάση του προσώπου και της ήρυδος των ματιών και των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε ποικίλους βαθμούς ασφάλειας. Το εμείς θα καταψηφίσουμε εν πάση περιπτώσει την έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Μπάτεν. Από τους μία γεγραμμένους για ένα λεπτό ο κύριος Κλάης. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σωστά Μιλάει ο εισηγητής για κάποια χαρακτηριστικά που σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με ε, τη συλλογή ε, ε, των στοιχείων, τη διατήρησή τους και τη σύγκρισή τους. Είναι καινούργια σχετικά διαδικασία. Και κάθε τρία χρόνια θα πρέπει να γίνεται σε βάθος αξιολόγηση και αποτίμηση. Και βεβαίως Χωρίς καμιά αμφιβολία υπάρχει κάποια εναρμόνιση στη διαχείριση των δεδομένων. Αλλά πάντα μια αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο ασθενής της κρίκος. Θεωρητικά θα πρέπει να έχουμε ενισχυμένη ε, φύλαξη των συνόρων, αλλά στην πραγματικότητα ε, έχει πολύ μεγάλες ελλείψεις και παραθυράκια ε, το σύστημα τα οποία εκμεταλλεύονται δίκτυα διεθνούς εγκληματικότητας και ε, κάνουν λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση ε, ανθρώπων και προωθούν τη λαθρομετανάστευση. Επιτέλους έχει έρθει η ώρα τα βιομετρικά στοιχεία να αξιοποιηθούν για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κλάις. Οι λοιποί ομιλητές τώρα. Για δύο λεπτά η κυρία Ντελάγκε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να απευθυνθώ το συνάδελφο μου Κοέγιο και να τον ευχαριστήσω. Κατάφερε σε πρώτη ανάγνωση να καταλήξει σε συμβιβασμό με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και την υποστηρίζω θερμά την πρόταση αυτή, ειδικά την αρχή που λέει ε, ένα πρόσωπο, ένα διαβατήριο. Αλλά θα πρέπει να βγω και σε λεπτομέρειε. Θα πρέπει αυτή η αρχή να προστατεύει τα παιδιά από τι απαγωγέ και τη διακίνηση. Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει δικό του διαβατήριο με ένα μικροτσίπ, έναν επαφικό πληθείο με τα βιομετρικά του στοιχεία. Και υπάρχουν χώρες που μέχρι τώρα εγγράφουν τα παιδιά στο διαβατήριο των γονέων. Στην Ολλανδία ε, κοστίζει το πολύ 48 ευρώ ε, ένα διαβατήριο και 8,5 για κάθε παιδί. Τώρα αν έχεις τρία παιδιά δηλαδή, ε, αντί για 120 ευρώ που κόστιζε πριν πρέπει να πληρώσει 240 ευρώ ως πενταμελής οικογένεια για τα διαβατήρια και των πέντε προσώπων. Και αυτό Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σημαντικό αν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών, αλλά αν κάποιο μπορεί να απαγάγει ένα παιδί, μπορεί να κλέψει και το διαβατήριό του εξίσου εύκολα. Και σε μερικέ περιπτώσει ακριβώ ε, δεν είναι μεγαλύτερη ασφάλεια όταν γράφεται το παιδί στο διαβατήριο του γονέα, που ξέρει ποιο γονέα αντιστοιχεί σε ποιο παιδί. Και τούμπαλιν θα πρέπει σε τρία χρόνια να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν χρειάζονται νέα μέτρα, νέα κανόνες για ε, τη διέλευση των συνόρων από παιδιά. Και ε, τότε ε, μόνο μπορούν να αρθούν οι διαφορές. Καλό και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει στην αξιολόγηση εάν και κατά πόσο αυτή η αρχή, το ένα πρόσωπο, ένα διαβατήριο οδήγησε στη μείωση των απαγωγών παιδιών. Γιατί αν η σημερινή συμβαστική πρόταση επέτυχε ή αν έχει ε, ανεπιθύμητες παρενέργειες. Κύριε Επίτροπε, η ασφάλεια των παιδιών μας χρειάζεται μόνιμη επαγρύπνηση. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα. Αν είναι προς όφελος και συμφέρον των παιδιών μας μέσω πρόθεσμα να κάνουμε και άλλα βήματα, θα βρείτε τους χριστιανοδημοκράτες στο πλευρό σας χωρίς καμιά αμφιβολία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Νταλάνκια. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Λαμπρινίδης, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή επικράτηση της άποψης του κοινοβουλίου έναντι της ε, προσπάθειας του συμβουλίου να επιβάλει το βιομετρικό φακέλωμα εξάχρονων παιδιών ε, είναι μια νίκη επί της αρχής επί της θεμελιώδους αρχής ότι όταν μιλάμε για προσωπικά μας δεδομένα αυτά μπορούν να συλλέγονται μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο αναλογικό και φυσικά χρήσιμο να γίνει κάτι τέτοιο. μια αρχή που τα τελευταία χρόνια φοβάμαι το συμβούλιο και η επιτροπή συχνά αγνοούν στι νομοθετικέ του πρωτοβουλίε. στην περίπτωση των ε, διαβατηρίων και των δαχτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών είναι προφανέ ότι τα παιδιά χρειάζονται δικά του διαβατήρια και δικά του γεωμετρικά στοιχεία σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε τι απαγωγέ την παιδική πορνογραφία ε, να αποτρέψουμε την εμπορία των παιδιών. ταυτόχρονα όμω είναι παράνομο προφανώ να συλλέγονται αυτά τα στοιχεία εάν δεν είναι απαραίτητα και όσον αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι για παιδιά έξι χρονών δεν είναι καν χρήσιμα αλλάζουν τα αποτυπώματα τόσο γρήγορα που τη διαβατήρια και η αναγνώριση μέσω αυτών καθίσταται άχρηστη. το κοινοβούλιο λοιπόν σήμερα πέτυχε την ισορροπία. απαιτεί από την επιτροπή μια σοβαρή μελέτη για να δούμε πραγματικά πότε μπορούν να έχουν προστασία τα παιδιά από τα δακτυλικά αποτυπώματα και επιτρέπει τη συλλογή τους μόνο για ηλικίες που ξέρουμε με βεβαιότητα ότι αυτό ισχύει τέλος σε κάθε περίπτωση για βιομετρικά στοιχεία διαβατηρίων ναι για την αναγνώριση του κατόχου τους ναι για την ταυτοποίησή του ναι για την εξακρίβωση ότι το διαβατήριο δεν είναι πλαστό όχι για τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακελώματος εκατομμυρίων αθώων πολιτών. ευχαριστώ. ευχαριστώ κύριε λαμπρινίδη. για ένα λεπτό το λόγο Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Η νέα κυκλοφορία των ε, διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία έρχεται να απαντήσει ε, στο πρόβλημα της πλαστογράφησης των διαβατηρίων της τρομοκρατίας και της λαθρομετανάστευσης. Γι' αυτό θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι αξιόπιστα τα στοιχεία και η συλλογή τους ακριβώς και να υπάρχουν κοινοί κανόνες που να τηρούνται από όλους βασικοί κανόνες για τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων που να εγγυώνται και την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Εγώ συμφωνώ με την τροπολογία ε, του εισηγητή να αναλυθούν οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών για να υπάρχει ασφάλεια στα έγγραφα. Ε, είναι σημαντικό ε, αυτό. Είναι σημαντικά τα βιομετρικά στοιχεία και ασφάλειά τους περισσότερο από το ίδιο το διαβατήριο. Υπάρχουν ε, τα βασικά έγγραφα όμως που μπορούν να πλαστογραφηθούν και αυτά. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Ρογκάλσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εναρμόνιση των στοιχείων για ασφαλείας και των χαρακτηριστικών ασφαλείας και των βιομετρικών για την ταυτοποίηση των προσώπων είναι κάτι το θετικό. Έτσι θα μπορούν να ελέγχονται καλύτερα τα έγγραφα, τα ταξιδιωτικά και καταπολεμεί την πλαστογραφία. Έχουμε την εγγύηση ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, τη λαθρομετανάστευση και την τρομοκρατία με τρόπο πιο αποτελεσματικό. Δεν υπάρχουν βέβαια δοκιμέ ακόμα για το πώς χρησιμοποιούμε τη νέα τεχνολογία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει το καθένα να έχει τους δικούς του κανόνες για την προστασία των πολιτών. Ας πούμε για το όριο ηλικία, Από ποια ηλικία και μετά θα πρέπει τα παιδιά να διαθέτουν διαβατήριο. Δεν επιτρέπεται να έχουμε ένα συλλογικό διαβατήριο για γονεί και παιδιά χωρί βιομετρικά στοιχεία. Θα πρέπει να είναι σε θέση ο ελεκτή να εξακριβώνει την ταυτότητα και των ανηλίκων. Κάθε πρόσωπο να έχει το δικό του διαβατήριο, έστω και τα παιδιά, να μην είναι με του γονεί στο ίδιο. Είναι σημαντικό και έτσι προστατεύεται και ο κάτοχος του διαβατηρίου ή των άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Θα πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί στη συλλογή και την τήρηση των στοιχείων. Ευχαριστώ κύριο Σαδάμου παρακαλώ είναι γεγονό ότι ο τροποποιητικό κανονισμό τον οποίο καλούμαστε να εγκρίνουμε ίσω επιφέρει βελτίωση σε δύο τρία κράτη μέλη όπου σήμερα λαμβάνονται τα βιομετρικά στοιχεία ακόμη και νηπίων και προσωρινά θα αποτρέψει κράτη μέλη από το να σύρουν σε λόγω διαδικασίε άτομα κάτω των δώδεκα ετών. Που βέβαια έτσι κι αλλιώ σημειώνουμε στο παρόν στάδιο σε κάποιε χώρε δεν είναι αναγκασμένα να ταξιδεύουν με προσωπικό διαβατήριο. Τι εξαιρέσει που προτείνονται πρέπει να τι αξιολογήσουμε βάσει των πραγματικών κινήτρων καθιέρωσή του αφού ανεξάρτητα του ηλικιακού ορίου λήψη βιομετρικών κάποια στιγμή όλοι ανεξαιρέτω μπορεί να βρεθούμε φακελωμένοι. Με τέτοιου κανονισμού επί τη ουσία συντηρείται και θεσμοθετείται ακόμη περισσότερο η χρήση μέθοδων φακελώματο, των απανταχού, πόσο μάλλον αθώων πολιτών και παραχωρείται το δικαίωμα τη διακίνηση ευαίσθητων προσωπικών μα δεδομένων. Είναι καθήκον μα λοιπόν να υπενθυμίσουμε στου πολίτε από του οποίου σε λίγου μήνε θα ζητήσουμε να ανανεώσουν την ψήφο του υπεραρχών και πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τέτοια μέτρα εμά δεν μα βρίσκουν σύμφωνου. Ευχαριστώ. Η καταγραφή των βιομετρικών δεδομένων είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί και το οργανωμένο έγκλημα και ε, μπορεί να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Αλλά πρέπει να είναι ε, σαφές ότι και η Frontex πρέπει να αναβαθμιστεί και με προσωπικό και μέσα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει σωστά τα καθήκοντά της. Εφόσον δεν υπάρχουν πλέον εσωτερικά σύνορα πρέπει να προστατεύονται επαρκώ τα εξωτερικά σύνορα. Υπάρχει και η υποψία και η είδηση ότι έχουν πλαστογραφηθεί με και ακόμη και δακτυλικά αποτυπώματα σε, ορισμένα, σε ορισμένες γερμανικές αρχές. Είναι σαφές πάντως ότι με την χρήση βιομετρικών δεδομένων πρέπει για τον απλό πολίτη να είναι εγγυημένη η προστασία των προσωπικών αυτών δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Μέλτσερ. Για δύο λεπτά η κυρία Μπάουερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Κοέλιο για την εξαιρετική έκθεση που συνέταξε επιθυμώ να τοποθετηθώ επί ορισμένων θεμάτων. Οι πρόσφατες εμπειρίες δείχνουν ότι το, το ε, σωματεμπόριο και κυρίως παιδιών έχει λάβει πλέον τρομακτικές διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αλλού. Γι' αυτό σημαίνει για μένα μια πρόοδο τα ανήλικα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να διέλθουν τα σύνορα μονάχα με δικό τους διαβατήριο. Αυτό προσφέρει ασφάλεια σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τον κίνδυνο της σωματεμπορίας. Από την άλλη μεριά, ως κάτοχος δικού του προσωπικού διαβατηρίου, το παιδί μπορεί να διέθεται σύνορα συνοδευόμενο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι θα πρέπει το διαβατήριο αυτό να περιλαμβάνει όχι μόνο τα ε, προσωπικά δεδομένα του παιδιού, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα του υπεύθυνου προσώπου που το συνοδεύει. Ε, η ε, έκθεση απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει έκθεση. Σε αυτήν πρέπει να τεθεί και να συζητηθεί και αυτό το θέμα για την λήψη ιδιαίτερων μέτρων για την προστασία των παιδιών. Σίγουρα ε, αυτό που ανέφερα μπορεί να αποτελέσει μια δυνατότητα για το μέλλον. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες οργανώσεις όπως τον ΟΑΣΕ, όπως τον είπα το αρμοστή των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες όπως την Interpol για να κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των παιδιών διότι οι εμπειρίες καταδεικνύουν ότι όλο και περισσότερα παιδιά ε, πέφτουν θύματα του Διεθνούς Σωματεμπορίου. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Φράντσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ να ε, συγχαρώ τον Κάρλος Κουέλιο. Τον Σεπτέμβριο του 2004 το ενέκρινε κανονισμό το Συμβούλιο για τα βιομετρικά δεδομένα και ε, δείκτες. Τώρα είναι απαραίτητο να ληφθούν και νέα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το σωματεμπόριο παιδιών. Η χρήση ε, παιδιών Συγγνώμη, η χρήση διαβατηρίων για τα παιδιά στη βάση του ένα πρόσωπο, ένα διαβατήριο μπορεί να αποτελέσει πρόοδο. Στη χώρα μου, την Πορτογαλία, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από καιρό ε, λαμβάνονται τα δεκτυρικά αποτυπώματα για παιδιά άνω των 6 ετών και αυτό λοιπόν έγινε ε, εύκολα μπορεί να γίνει εύκολα δεκτό από το πορτογαλικό κοινό. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες μέλη, όπως η Πορτογαλία, που έχουν ένα κατόφλιο ηλικία 6 ετών για την λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και ε, επιτρέπει η οδηγία να μην τροποποιήσουν την εθνική του νομοθεσία. Δεν είναι όμω μόνο το θέμα των ε, διαβατηρίων. Στα διαβατήρια ενδιαφέρει το επίπεδο ασφάλειας. Αλλά πρέπει να είναι το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλεια και των εγγράφων τα οποία χρησιμοποιούνται για την έκδοση των διαβατηρίων. Η έκθεση λοιπόν κάνει ένα βήμα παραπέρα για την εγγύηση των προσωπικών δεδομένων των ε, ενδιαφέρον προσώπων. Σας ευχαριστώ κύριε Φράντσα. Ο κύριος Μπρέιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω την εισήγηση του κυρίου Κοέλιο που έκανε τη δουλειά του με εξαίρετο τρόπο όπως ο συνήθως. Σύμφωνα επίσης με τις προτάσεις που ακούσαμε σήμερα, κυρίως για την αρχή ένα άτομο, ένα διαβατήριο, αλλά θα ήθελα να ακούσω την απάντηση στην ακόλουθη ερώτηση από την Κομισιόν και ίσως από τον εισηγητή. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση των παιδιών που ταξιδεύουν μόνα τους χωρίς να συνοδεύονται, διότι δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική για τα έγγραφα με τα οποία πρέπει να ταξιδεύει ένα τέτοιο παιδί. Σύμφωνα με την έκθεση, το έγγραφο θα πρέπει να αναφέρει το άτομο που έχει την γονική ευθύνη για το παιδί, αλλά πολύ συχνά το παιδί ε, ταξιδεύει συνοδευόμενο από άλλα μέλη της οικογένειας, ακόμα και με άτομα που δεν έχουν γονική ευθύνη πάνω στο παιδί. Υπάρχει επίσης ε, κάτι άλλο που με ενοχλεί. Όντως, πώς θα μπορέσουμε να αφήσουμε ένα παιδί 6 ετών να ταξιδεύει μόνο του με το αεροπλάνο, εντάξει, αλλά ας αφήσουμε ε, τα τραύματα που μπορούν να δημιουργηθούν για ένα τέτοιο παιδί που ταξιδεύει μόνο του και ε, που ε, παραδίδεται σε κάποιον που τον περιμένει στο αεροδρόμιο της άφηξης, αλλά στην περίπτωση ενός ταξιδιού με τρένο ή με λεωφορείο ενός παιδιού, τι πρέπει να γίνει αν οι γονεί δεν είναι τόσο ανεύθυνοι ώστε να στέλνουν τα παιδιά τους μόνα τους να ταξιδεύουν με τρένο ή λεωφορείο ε, σε χαμηλή ηλικία. Το, εκεί πρέπει να διαρωτηθούμε τι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ε, θαραλέοι ε, σχετικά με τις θέσεις μας για το θέμα αυτό και σχετικά με την ασφάλεια την ασφάλεια των πηγών, των εγγράφων πηγών για την έκδοση των θεωρήσεων διαρωτώμαν. Υπάρχουν συστήματα στις χώρες μας που επιτρέπουν απάτες και καταχρήσεις στην περίπτωση έκδοσης θεωρήσεων και ταξιδιωτικών εγγράφων. Και ακόμη μια ερώτηση για τον εισηγητή. Τι πρέπει να γίνει όταν ένα άτομο βρίσκεται ε, στο σύνορο και όταν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του ταξιδιωτικού του εγγράφου δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία της βάσης των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Κάστεν Κλέρκ. κύριε και κύριοι, χιλιάδες παιδιά πέφτουν κάθε χρόνο θύματα του σωματεμπορίου και ακόμα περισσότερα απαγωγών κυρίω ανήλικα παιδιά. Γι' αυτό χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τροποποίησή τη του παλαιού κανονισμού λαμβάνει υπόψη τα θέματα αυτά. Ζητούμε από κάποια ηλικία και μετά τα παιδιά να έχουν διαβατήρια τα οποία να περιλαμβάνουν τα προσωπικά του δεδομένα. Αλλά αυτό το κάνουμε μόνο για να προστατευτούν καλύτερα τα παιδιά. Και η προστασία μπορεί να είναι καλύτερα εξασφαλισμένη εφόσον το παιδί έχει δικό του διαβατήριο με τα βιομετρικά του δεδομένα και εφόσον σε αυτό περιλαμβάνονται και τα ονόματα των προσώπων που έχουν την ε, ευθύνη για το παιδί αυτή. αυτό. Πρέπει να είναι εξασφαλισμένη ωστόσο η χρήση των βιομετρικών διαδεδομένων και να είναι εγγυημένη η ασφαλειά τους και πρέπει να είναι ανα πάσα στιγμή δυνατό να ε, διευκρινιστεί ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. Και πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι κατά της κατάχρησης δεδομένων. Έχω μια καταρχήν εμπιστοσύνη στις ε, κρατικές αρχές της ε, χώρας μου, αντιθέτως από ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για να τα εμπορεύονται με, με, άλλες. Γι' αυτό οι αρχές ελέγχου πρέπει να είναι κρατικές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίθετα από ό,τι συμβαίνει εδώ θα πρέπει να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις και να λάβει υπόψη την άποψη του ε, ε, εντεταλμένου τα προσωπικά, την προσέγγιση προσωπικών δεδομένων και συνεχίζει στα πορτογαλικά συγχαίροντας τον κύριο Κοέλιο για την εργασία του. Ευχαριστώ κύριε Κράσιλντορφλερ. Το λόγο έχει για δύο λεπτά τώρα η κυρία Στράφκοβα. Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ με τη σειρά μου τον εισηγητή κύριο Κοέγιο για την ισορροπία που κατάφερε να βρει στην έκθεσή του. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε διάφορα έγγραφα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές αναπροσαρμογές που χρειάζονται για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, της λαθρομετανάστευσης ε, και της διακίνησης ανθρώπων. Για τι φτωχέ χώρε όπως είναι η Βουλγαρία ε, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι νέε προδιαγραφές και πόσο σημαντικές θα είναι για την προστασία των εξωτερικών συνόρων τη Ένωση από τα φαινόμενα αυτά. Έχουμε ε, ανηλίκους που ε, έχουν εξαφανιστεί και αγνοούνται χωρίς καμία πληροφόρηση. Και τώρα ε, νομίζω θα αυξηθεί η ασφάλεια και οι προδιαγραφές για τον έλεγχο των καταστάσεων αυτό ακόμα και στα διαβατήρια των πιο νεαρών πολιτών, των ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ταξιδεύουν είναι εκτός της Ένωσης. Οι πληροφορίες για τα στοιχεία ανηλίκων ε, μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε τη διακίνησή τους. Το trafficking. Υπάρχει το θέμα της ελεύθερης διακίνησης και των οικογενειών που θέλουν να ταξιδεύουν με μικρά παιδιά. Και δεν θα πρέπει αυτό να εμποδίζεται από το υψηλό κόστος διαβατηρίων για τα τέκνα τους. Θα ήθελα λοιπόν τέλος να Απευθύνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη να μην είναι απαγορευτικές διατάξει για να μπορούν να ταξιδεύουν ακόμα και τα παιδιά στην Ένωση. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Γκραβόφσκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον εισηγητή και να του πω ότι υποστηρίζω την έκθεσή του, την οποία θεωρώ σημαντική και καλή. Το διαβατήριο είναι έγγραφο το οποίο εκδίδει κάθε χώρα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής της νομοθεσίας. Είναι διαφορετικά διαβατήρια με το ίδιο εξώφυλλο. Χρειάζεται όμως να βρούμε και μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης ασφάλειας του εγγράφου αυτού και της ανάγκης ταυτότητας, ταυτοποίησης των πολιτών αλλά και των προσώπων που εισέρχονται από αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα πρέπει να μας δίνει τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε ε, το οργανωμένο έγκλημα που χρησιμοποιεί ε, παραχαραγμένα διαβατήρια, όπως ε, επίσης το σωματεμπόριο παιδιών κλπ. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη η έκθεση. Τίποτε δεν δείχνει ότι τα όσα ζητούμε τώρα για τα διαβατήρια οδηγούν σε περιορισμούς ε, στις χώρες μέλη ό,τι αφορά την δυνατότητα έκδοσης διαβατήριων. Επισημαίνω την αρχή ένα πρόσωπο, ένα διαβατήριο, με την οποία είμαι σύμφωνη. Είναι καλό για τα παιδιά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, επιτρέψουμε να οδηγήσει σε οικονομικές δυσχέρειες των οικογενειών εκείνων οι οποίες θέλουν να εκδώσουν διαβατήρια για τα παιδιά τους αλλά ε, μπορεί να μην έχουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα. Ε, να αναφέρομαι και στο γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια αναθεώρηση σε μια τριετία. Απευθύνω έκκληση και για το ότι θα πρέπει ο ρόλος του Ευρωπαίου εντεταλμένου την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να γίνει διαβούλευση μαζί του για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Γραμπόσκα. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό ο κύριος Εβαντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Κουέλιο. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή για τους 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρώπης ε, για την ασφαλειά τους και για τα αντιτρομοκρατικά μέτρα. Αν υπάρχει η τεχνολογία όπως λέχθηκε θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά στα παιδιά Αντζελίλη και ο κύριος Λαμπρινίδης ε, είπε ότι μπορεί να είναι ζωτικό όπλο κατά ε, της εμπορίας των παιδιών. Αλλά νομίζω ότι το νέο άρθρο 3 είναι το καλύτερο, ότι ο σκοπός δεν είναι να εξακριβώσουμε την γνησιότητα ενός εγγράφου, αλλά ε, την ταυτότητα του κατόχου με συγκρίσιμα στοιχεία αξιόπιστα. Οι περισσότερα, περισσότερες χώρες βασίζονται σε φωτογραφίες, αλλά κανείς, ούτε εσείς κύριε Πρόεδρο, το κύριο Μπαρόσο, δεν μοιάζεται με την φωτογραφία του διαβατηρίου σας, ούτε κανείς δεν θέλει και να μοιάζει. Υπάρχουν λοιπόν νέες διαδικασίες, νέες μεθόδοι, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπε η κυρία Γκάσεκ, ο κύριος και άλλοι που δεν βρίσκονται εδώ την αντιβρετανικές τους συμβολές. Το σύστημα ίσως του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι καλύτερο ούτε χειρότερο από άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως έχουμε τα υπέρ και τα κατά, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι με τεχνολογία που θα υπάρξει πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και όπως είπε η κυρία Γκραμπόσκα θα πρέπει να τροποποιούμε, να προσαρμόζουμε συνεχώς χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα τα μέσα που μας παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ακολουθούν τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές. για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Ε, η προστασία των παιδιών και των ανηλίκων από το λαθρεμπόριο χρειάζεται ε, ακριβώς και απαιτεί το να έχει κάθε παιδί το δικό του διαβατήριο. Και κλείνει το μικρόφωνο ο μιλητής. Excuse me once more. Έλεγα λοιπόν ότι η προστασία των παιδιών απαιτεί τα παιδιά να έχει ναι, το καθένα το δικό του διαβατήριο, κάθε πρόσωπο να έχει διαβατήριο. Δηλαδή, κάθε ε, ανήλικος που ταξιδεύει πέρα από τη ζώνη Σέγγεν θα πρέπει να έχει ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό απλουστεύει τους ελέγχους στα σύνορα. Υπάρχει επίσης και μια τηλεφωνική γραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ανηλίκων, για τις καταγγελίες για παιδιά που τη χάνουν σεξουαλικής κακοποίησης, ε, κακομεταχείρισης ή ε, απαγωγής. Ε, είναι επίσης ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των βιομετρικών στοιχείων. Σίγουρα και το κατανοώ θα πρέπει να αναλύσουμε τις αδυναμίες, τα προβλήματα ταυτοποίησης βάσει δακτυλικών αποτυπωμάτων των αλληλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση και σύστημα. Ε, κοπά για ένα λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και εγώ τον Κάρλος Κοέγιο, ε, να καλωσορίσω την πρωτοβουλία του. Είναι πραγματική πρόοδος μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης γίνεται η σύνδεση μεταξύ του ταξιδιωτικού εγγράφου και του κατόχου του και εισάγεται η αρχή ένα πρόσωπο, ένα διαβατήριο, ένα ταξιδιωτικό έγγραφο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξή τρία στοιχεία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε ποιε είναι οι αρχέ αλλά και οι εξαιρέσει που προβλέπει η έκθεση για την πρακτική εφαρμογή των προτάσεων. Δηλαδή θα πρέπει ε, ακριβώς μετά από μία τριετία να αναθεωρηθεί και να αναλυθεί η κατάσταση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουν τι συστάσεις πρέπει να γίνουν ε, και ποιες είναι οι θεωρητικές αρχές και ποια είναι η εφαρμογή τους στην πράξη ε, και ποια τα εμπόδια. Άλλο πρόβλημα, δεύτερο, έχει να κάνει με την ασφάλεια των δεδομένων που φυλάσσονται και τηρούνται και η προστασία ε, της προσωπικής ζωής του κατόχου του διαβατηρίου. Και τρίτο, θα ήθελα να σας πω ότι χρειάζονται κοινέ αρχές και κανόνες για τα ταξιδιωτικά έγγραφα, για τα διαβατήρια. Είναι απόλυτα απαραίτητο αυτό για να υπάρχει ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων και να μην έχουμε πλαστογραφίες. Ευχαριστώ κύριε Πόπα. Για ένα λεπτό το λόγο έχει τώρα η κυρία Ρούρ. Euh, άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω κύριε Κοέλιο και είναι μεγάλη χαρά που εργαστήκαμε μαζί σας διότι επιδεικνύεται μεγάλη αρμοδιότητα, έχετε μεγάλη ικανότητα να ακούτε τους άλλους, να αναλύετε τα θέματα και χάρη σε εσάς καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Κοέλιο, Σηκωθείτε σας παρακαλώ και κάντε καμιά υπόκληση εδώ. Πολύ ωραία. Για ένα λεπτό το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Η Ρουμανία την 1η Ιανουαρίου ε, υιοθέτησε τα βιομετρικά διαβατήρια με 50 στοιχεία ασφαλείας και για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, ταυτοποίηση και του προσώπου και των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Έχει κάνει πολύ σημαντικό βήμα η Ρουμανία προς το σύστημα και το χώρο Σέγγεν που θα ενταχθεί το 2011. Αυτό το νέο βιομετρικό διαβατήριο ε, εξαλείφει και τις τελευταίες επιφυλάξεις για την άρση θεώρησης ε, visa waiver των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν αντικειμενικά λοιπόν στοιχεία στη διάθεσή τους πλέον και, ε, μόνο υποκειμενικά είναι εκείνα τα εμπόδια που ε, αντικρούν την άρση των θεωρήσεων. Για ένα λεπτό, η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή με τη σειρά μου. Η ευρωπαϊκή εναρμόνιση των ε, προδιαγραφών ασφαλείας και των βιομετρικών διαβατηρίων ε, αντιπροσωπεύει ε, τη διεύρυνση του κεκτημένου του Σέγγεν. Πρόκειται για ένα ανεπαφικό πλυνθείο στο ε, διαβατήριο ένα τσίπ, δηλαδή που δεν χρειάζεται ε, επαφή. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να σέβονται τις κοινοτικές ρυθμίσεις ε, για την προστασία δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων και αυτό να το εγγυάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στα σύνορα αλλά και στη βάση των δεδομένων εφόσον αυτό το προβλέπει η Εθνική Νομοθεσία. Θα ήθελα να συμπιστήσω την προσοχή στο γεγονό ότι ένα βιομετρικό διαβατήριο για κάποιον που δεν μπορεί να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα ε, δυσκολεύει τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Ματσάκης παρακαλώ. Πρόεδρε. Κανένα νομοταγή πολίτη δεν θα πρέπει κανονικά να ανησυχεί για την ταυτότητά του ή το παιδιών του. Γι' αυτό καλωσορίζω τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων στα δημόσια ταξιδιωτικά έγγραφα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξή μόνο για μελλοντική αναφορά. Είναι γεγονό ότι δεν υπάρχουν βιομετρικά χαρακτηριστικά που να παραμένουν ατόφια και γνήσια ε, από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλίκη εκτό από ένα, το αποτύπωμα DNA. Το δακτυλικό αποτύπωμα και μετά θάνατον ακόμα. Και μπορεί ε, ε, κανένα σήμερα να ταυτοποιηθεί χρόνια ολόκληρα μετά ε, από το θάνατό του αν υπάρχει έστω και ψήγμα των οστών του που έχουν απομείνει. Είναι λοιπόν το γενετικό αποτύπωμα, είναι γρήγορη μέθοδος, φτηνή και χρειάζονται λίγα μόνο κύτταρα. Ή, αρκεί κανείς να πάρει λίγο υλικό από το πλενογόνο το στοματικό ε, ή ε, κάποιο άλλο κυταρικό υλικό για να το διαπιστώσει. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε το αποτύπωμα το γενετικό, όχι το δακτυλικό πλέον, το DNA. Θα μπορούσε να είναι και ένα βιομετρικό στοιχείο και το μόνο που εγγυημένα παραμένει το ίδιο για κάθε ε, πολίτη και για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ματσάκη. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Πίρκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κοέλιο και με την ευκαιρία το συγχαίρω κιόλα εξαιρετική ποιότητα η έκθεση που ακολουθεί την ποιότητα και άλλων εκθέσεων του κ. Κοέλιο Και εξ αρχή ο κ. Κοέλιο είπε ότι ο στόχος του είναι η επίτευξη της ασφάλειας των παιδιών, η οποία βέβαια ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί με καλύτερο εξοπλισμό, με ε, συγκεκριμένα με την ε, ε, λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων που επιτρέπει την ταυτοποίηση του παιδιού εφόσον διαβαίνει τα σύνορα. Είναι λοιπόν ένας στόχος για την επίτευξη ασφάλειας των παιδιών. Τώρα, εάν θα είναι 6 χρονών ή 12 χρονών, αυτά ας τα διευκρινίσουν οι τεχνικοί. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να ληφθούν κτηρικά αποτυπώματα ήδη από τις ηλικίες των 6 ετών εφόσον πρόκειται για την ασφάλεια του ίδιου του παιδιού. Βεβαίω και πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά και οι διατάξει για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Είναι καθήκον του κράτου μέλου. Εάν όμω έχουμε εν τέλει ασφαλή διαβατήρια και τηρούνται και οι διατάξει για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τότε θα έχει κάνει πια η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό για το συμφέρον των παιδιών και κατά του σωματεμπορίου ε, παιδιών. Ευχαριστώ. κύριο Μπάρο. Eh Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι όλη αυτή η συνέλευση απέτησε φοροτιμή στην εργασία του κύριου Κοέλιο και στα προσόντα του και ε, συμμερίζομαι και εγώ την άποψη της κυρίας Ρούρα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω ε, και ας επαναλάβω τα λόγια του Προέδρου Γεράρντ Πρέ, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστες και συγκρίσιμα ε, στοιχεία βιομετρικά. Γι' αυτό έχουμε αυτό το ραντεβού το οποίο προβλέπετε που θα μας επιτρέψει να κάνουμε μια καλύτερη χρήση των πιο προχωρημένων τεχνολογιών για να εξασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια σε αυτόν τον χώρο ελευθερίας στον οποίο βρισκόμαστε. Και χαίρομαι λοιπόν που βλέπω το Κοινοβούλιο τόσο ε, δεσμευμένο για αυτόν τον χώρο για να είναι πιο ασφαλής η παρουσία και η μετακίνηση των παιδιών. Με ρωτήσαν αν έχουμε ήδη την απόδειξη ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των διαδικασιών ταυτοποίησης υπάρχει. Θα έλεγα ότι μόνο η χρήση εφαρμογή θα μας επιτρέψει να εξακριβώσουμε την αποτελεσματικότητα. Αλλά απριόρι νομίζω ότι μια καλύτερη ταυτοποίηση των παιδιών που ταξιδεύουν μόνα τους θα μας δώσει περισσότερη ασφάλεια. Πάντως δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη αυτό το βασικό στόχο. Θα ήθελα να δώσω μερικές απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις Πρώτα απ' όλα να επαναλάβω να υπογραμμίσω ότι πάντοτε τονίσαμε το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Ο ελεγκτής της προστασίας των δεδομένων ερωτήθηκε για την βασική πρόταση, υπέβαλε παρατηρήσεις που λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι σε σχέση ε, με τα άτομα που πρέπει να ταυτοποιηθούν. Υπάρχει εναρμόνιση των προτύπων μας με, τον, με την, ε, την, οργάνωση, την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Και αυτό θα παρακινήσει το διάλογο με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι για τα διαβατήρια των παιδιών βεβαίως υπάρχει μια οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες, αλλά αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Για να ταξιδέψει ε, κανείς ε, στο χώρο Σέγγεν απαιτείται μόνο η ταυτότητα. Το διαβατήριο απαιτείται για τα ταξίδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω και να επιβεβαιώσω ότι η Κομισιόν θα κάνει μια μελέτη συγκριτική των υφισταμένων κανόνων στα κρατημέλη σχετικά με τα ταξίδια των ανηλίκων παιδιών που ταξιδεύουν μόνα τους και θα προτείνουμε εν ευθέτω χρόνο στο Συμβούλιο να λάβει τα μέτρα που επιβάλλονται για μια καλύτερη προστασία των παιδιών και ε, για την καταπολέμηση της εμπορίας των παιδιών. Βεβαίως το Κοινοβούλιο θέλει μια τέτοια μελέτη και εγώ αναλαμβάνω να μεριμνήσω ούτω ώστε οι υπηρεσίε μου να εκπονήσουν αυτήν την μελέτη το συντομότερο δυνατόν και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ευχαριστώ άλλη μια φορά το Κοινοβούλιο για την επικοδομητική συμβολή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής, ε, κύριος Κόγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν είναι ένα το συμπέρασμα της συζήτησης, αυτό είναι το εξής. Κατά πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο εκφράζεται μια ανησυχία. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διακίνηση προσώπων, κυρίως το θέμα των παιδιών. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο. Σχεδόν όλοι οι προλαλήσεντες αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους σκιώδεις ηγητές για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ την κυρία Ρου για τα καλά σας λόγια, αλλά και η δική σας συνεργασία ήταν πάρα πολύ πολύτιμη για να καταλήξουμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο κύριο Μπαρό και τη Γαλλική Προεδρία. Σας ευχαριστώ όλους σας που συμφωνείτε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση της εμπορίου παιδιών. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Ε, η αξιοπιστία των δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών σε λεγόμενα έγγραφα breeder που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων εγγράφων και άλλα τεχνικά ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, κάποιος ρώτησε αν υπάρχει δυνατότητα για μας να πούμε ότι είναι ασφαλή τα διαβατήριά μας. Για να είμαι ειλικρινής, Πρέπει να σας πω ότι αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες που έχουν πιο ασφαλή διαβατήρια και κάποιες άλλες λιγότερο. Γι' αυτό χρειάζεται και εναρμόνιση στα βασικά έγγραφα, τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ταξιδιωτικών εγγράφων. Αλλά εκεί σας είπα η αρμοδιότητα δεν είναι κοινοτική, παραμένει κρατική αρμοδιότητα η έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Ελπίζω εδώ να είναι καλή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα κείμενα Breeder το θέμα δεν έχει νόημα να έχουμε ασφαλέστερα ταξιδιωτικά έγγραφα και διαβατήρια εάν αυτά υπονομεύονται κατά την έκδοσή τους. Και βέβαια ε, είναι θέμα κρατικής αρμοδιότητας, αλλά καλό είναι να ενταλλάσσουμε και βέλτιστες πρακτικές και το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο να σημαίνει ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόηγιο. Ολοκληρώνεται εδώ το σημείο αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ε, και τώρα ακολουθεί η έκθεση του κυρίου Καπάτο με θέμα την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Καπάτο ε, για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.